επιτροπές για να μην συνηθίζουν και προσιλώνονται σε ένα μονάχα είδος αίθουσας και αυτό βοηθάει την ποικιλία της εργασίας των επιτροπών. Καλώς ήλθατε λοιπόν σε αυτή την στρογγυλή τράπεζα που θυμίζει τον βασιλέα Αρθούρο και τους υπότες του στο Κάμελοτ. Εγώ σας βλέπω, δεν σας βλέπω στην άκρη του ορίζοντα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Έχετε το σχέδιο μέσα στη διάταξη μπροστά σα. Έχετε κάποιε παρατηρήσει σχετικά. Εάν έχει ούτω, μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά 18-14 Φεβρουαρίου 2013. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Και έχουμε μετά την πληροφόρηση για τους τριμερείς διαλόγους. Μου είπαν την επόμενη φορά θα πρέπει να έρθουμε στο θέμα αυτό. Υπηρεσίε εδάφους τέσσερα Ο κύριο Ζασάντα είναι παρόν, θα του δώσω και τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω όλους τους χειώδεις συζητητές για τις πολλαπλές συναντήσεις που είχαμε μέχρι στιγμής για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, τις τροπολογίες συγκεκριμένα και να καταλήξουμε σε 10 περίπου συμβιβαστικές τροπολογίες. Έχουμε ξεκινήσει να εργαζόμαστε για το θέμα αυτό εδώ και ένα χρόνο περίπου και νομίζω ότι είμαστε πια πολύ κοντά στην ε, κατάληξη των εργασιών μας που θα είναι η αυριανή ψηφοφορία. Φυσικά είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν ικανοποιημένοι με το τελικό αποτέλεσμα, αλλά θέλω να σα υπενθυμίσω ότι θα λάβει χώρα και μια ψηφοφορία στην Ολομέλεια, η οποία θα συμπληρώσει την πρώτη ανάγνωση του θέματος αυτού και συνέχεια έχουμε την δεύτερη ανάγνωση αφού έχουμε και την άποψη του Συμβουλίου ενδιαμέσως. Αυτό το οποίο εγώ έχω συμπεράνει μετά από ένα έτος εργασίας είναι ότι έμαθα την πιο συνηθισμένη λέξη που λέγεται στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι η λέξη οδηγία, η λέξη τροπολογία, η λέξη πολιτική ομάδα. Είναι η λέξη συμβιβασμό. Αλλά είναι μια καλή λέξη, δεν είναι κακή λέξη ο συμβιβασμό. Εάν δεν είναι κανεί ποτέ ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα και βγαίνουν όλοι από την αίθουσα συνεδριάσεων λέγοντας ότι η λύση την οποία πετύχαμε δεν είναι τέλεια αλλά είναι ανεκτή, είναι επαρκή. τότε έχουμε πετύχει μια σωστή συμβαστική λύση και νομίζω ότι αυτό έχουμε καταφέρει να πετύχουμε μεταξύ μα εκτό από ένα θέμα που έχει να κάνει με την συμβαστική λύση H λατινικό που έχουμε δύο εκδοχέ του κειμένου. Οι περισσότερε συμβαστικέ λύσει έχουν γίνει δεκτέ από όλου ή σχεδόν όλε τι πολιτικέ ομάδε, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι αξιοσημείωτο και είναι μια μεγάλη επιτυχία των διαπραγματεύσεων μα. στην ε, αξιολόγηση που κάνω των συζητήσεων, εκτιμώ ότι παρά το γεγονό ότι οι περισσότερες συζητήσεις περιστρεφόντουσαν για το αν θα πρέπει να έχουμε περαιτέρω φιλελευθερωποίηση με τρεις ή τέσσερις υπηρεσίες εξυπηρέτηση στα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι, σαφές, είναι σαφώς πιο σημαντικό στο έγγραφο είναι κάποια θέματα τα οποία έμειναν στο περιθώριο της συζήτησης, όπως η εισαγωγή μια κοινή διαδικασίας για υποβολές προσφορών για εξυπηρέτηση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Κάτι το οποίο να είναι σαφές και αναγνώσιμο για όλους, να μην υπάρχουν 27 χωριστέ διαδικασίες, αλλά μόνο μία διαδικασία. Επίσης, μία ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα αεροδρόμια και των 27 κράτων μέλων. Επομένω, ένα πάροχο υπηρεσιών εδάφου που θέλει να δώσει υπηρεσία σε 27 κράτη-μέλη, δεν θα είναι υποχρεωμένος να ζητά 27 εγκρίσεις. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν δεν ήταν καν στοιχείο της πρώτης Κομισιόν, είναι τα ελάχιστα πρότυπα. Τελικά λοιπόν, για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια θα θεσπιστούν κάποια πρότυπα τα οποία θα πρέπει να τηρούν όλοι. Και αν κάποιος πάροχος δεν τηρεί τα πρότυπα μπορεί να χάσει τη θέση του στο, ε, στο αεροδρόμιο αυτό ή μπορούν να του επιβληθούν κυρώσεις. Και κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους αυτούς που κατέθεσαν τροπολογίες. Πάνω από 500 τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στις διαπραγματεύσεις για τις συμβαστικές λύσεις και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που τις ενέκριναν και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Φλέκενστάιν, σοσιαλιστές. Μερσή κύριε Πρόεδρε. Πάντα μια συμβαστική λύση σημαίνει ότι όλα τα κομμάτια, όλες οι ψηφίδες έχουν έρθει στη θέση τους και φυσικά έχουμε όλοι κάνει μεγάλες προσπάθειες για να καταλήξουμε στις λύσεις αυτές και εσείς το ίδιο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι για την έννοια της υπεργολαβίας συγκεκριμένα <clears throat> για το τι ακριβώς είναι γενικού χαρακτήρα συμφωνία όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά σημεία και για όλους μας και σε ό,τι αφορά τα κατόφλια τα οποία είχατε προτείνει. Πιστεύω ότι η λύση που έχουμε επιτύχει κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επομένως, πιστεύω έχουμε μία σειρά από σημεία τα οποία θα μπορούσε και το Συμβουλίο να τα αποδεχτεί. Υπάρχουν κάποια σημεία όπου υπήρξαν αποκλήσεις απόψεων μετά υπήρξαν συμφωνίες, μετά πάλι διαφορές μεταξύ μας και αυτό ήταν τα θέματα που άπτονται της επικουρικότητος. Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικές ε, εκδοχές που θα πρέπει να ψηφίσουμε αύριο. Και εγώ από τη δική μου πολιτική ομάδα θεωρώ ότι αν γίνει δεκτή η δική μας πρόταση, η, τροπολογία, η συμβαστική τροπολογία λοιπόν των σοσιαλιστών, εάν γίνει δεκτή, θα <clears throat> υποστηρίξουμε στο τέλο και στη συνολική ψηφοφορία το πακέτο αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ, εκ μέρου των Φιλελευθέρων, νομίζω μιλάτε εκ μέρου του κυρίου Κλίντ. Πράγματι, ο κύριο ε, Κλίντ ε, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα εδώ. Είχε λυμμένε υποχρεώσει. Ευχαριστώ όμω πάρα πολύ για τη συνεργασία και για την επώδυνη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία που κράτησε και πολύ καιρό. Ούτε και αύριο μπορεί να έρθει. Τι να κάνουμε. <coughs> Μου είπε λοιπόν ότι η δική του εμπειρία αλλά και άλλων ε, συναδέλφων μήπως μιλά πολύ δυνατά. Όχι, είναι εντάξει. Λοιπόν, σε ορισμένα αεροδρόμια είναι δυνατόν να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις. Και χαίρεται πάρα πολύ, τουλάχιστον όσον αφορά τις ε, προδιαγραφές ε, και την πιστοποίηση, ακολουθείται η σωστή κατεύθυνση. Ε, το θέμα των παρόχων ότι αυτός ο αριθμός πρέπει να περιοριστεί. Κατά την άποψή του δεν είναι αυτό το μόνο κρίσιμο θέμα. Κατά τα άλλα, λέει ότι εξακολουθεί να είναι επιφυλακτικός όσον αφορά τις προτάσεις από την Επιτροπή Επασχόλησης. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι οι φιλελεύθεροι μιλήσαμε για το θέμα αυτό και τις σημαντικές προτάσεις του κυρίου Σασάλα τις θεωρούμε θετικές ε, γιατί έκανε πάρα πολλά, προσπάθησε να έρθει κοντά μας όσον αφορά τις προδιαγραφές, ε, τις υπεργολαβίες. Βεβαίως και έγινε λόγος ε, για την επικουρικότητα. Οι περισσότεροι είναι υπέρ αυτής, αλλά και όλοι οι άλλοι λένε ότι να υπάρχουν τρεις πάροχοι και μεταβατική περίοδος 10 ετών. Αυτό είναι αποδεκτό. Δηλαδή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ε, αυτή η λύση, για τους φιλεύθερους τουλάχιστον, είναι η καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, μας εξέπληξαν οι συζήτησεις ε, μέχρι στιγμής Υπάρχει μια ομάδα βουλευτών που μας μιλούν συνέχεια για την επωνομαζόμενη ενωσιακή μέθοδο. Όλα θα πρέπει να γίνονται τηρώντας αυτήν την μέθοδο. Λοιπόν, για αυτό το συγκεκριμένο φάκελο τι διαπιστώσαμε. Διαπιστώσαμε ότι τα εθνικά αντανακλαστικά υπερτέρησαν. Αυτό ισχύει για τις μεγάλες πολιτικές ομάδες ε, του Κοινοβουλίου. Μα εξέπληξε αυτό σε μεγάλο βαθμό ομολογουμένω. Δεύτερον, η συμβαστική 1. Έχουμε μελετήσει μακρόν αυτή την ε, συμβαστική πρόταση και τελικά αποφασίσαμε να την εγκρίνουμε διότι κάνουμε ένα έστω και μικρό βήμα προς την απελευθέρωση. Ακονίζουμε τα δόντια μας ε, χονδρικά και θα κάνουμε αυτή την υποχώρηση, θα υποστηρίξουμε τελικά την ε, συμβαστική πρόταση. Θα θέλαμε ταυτόχρονα να απευθύνουμε διάφορες ερωτήσεις προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά ζητήματα, παραδείγματο χάρη στην παράγραφο H. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει σχετικά με την πορεία των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε επικαιροποιημένε πληροφορίες. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο, όπως και η ομάδα μας, θα διαγράψει, θα καταργήσει όλα αυτά τα επίμαχα σημεία από την πρότασή της. Ιδανικά θα θέλαμε φυσικά να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Γνωρίζουμε όμως από πικρή πείρα ότι σπάνια ε, απαντά σε ερωτήσεις ο ε, εκάστοτε εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Επαναλαμβάνω ότι θα ε, υποστηρίξουμε την επίμαχη συμβαστική πρόταση γιατί θέλουμε πάση θυσία να προχωρήσει αυτή η πρόταση για την ναι, χορύπανση και τις χρονοθυρίδες έχουν ε, ληφθεί διάφορες αποφάσεις ε, αλλά στα πλαίσια ενός πάζα ρέματος για να κερδίσουμε άλλα στοιχεία της πρότασης ελπίζω ότι Αύριο θα καταλήξουμε σε μια τελική λύση. Περιμένουμε την απάντηση ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε, κύριο Κράμερ. Ε, η κυρία Λίχτενμπεργκ δυστυχώ έχει καθυστερήσει, έχει καθυστερήσει πτήση τη και γι' αυτό θα μιλήσω εξ ονόματό τη. Ε, καταρχήν θέλω να πω ότι είναι πολύ αρνητικό για το Κοινοβούλιο όλο αυτό που συμβαίνει. Ε, συζητήσαμε διαμακρών και λήφθη η απόφαση με μία μόνο ψήφο. Στην Ολομέλη όμως αναπέμφθηκε το θέμα με συντηρητική πλειοψηφία και τι κάνουμε, ε, το ξανασυζητάμε. Αυτό για μένα δεν είναι και βουλευτισμό. Είχαμε καταλήξει μία θέση και θα έπρεπε το Κοινοβούλιο, μάλλον συγγνώμη το Συμβούλιο να έρθει προ τη δική μα την πλευρά. Ε, Τώρα λοιπόν έχει κατατεθεί μια νέα πρόταση που προβλέπεται μεταβατική περίοδο 10 ετών. Αυτό και μόνο δείχνει, μιλάει από μόνο του πόσο επίγονε το θέμα. Και αν ε, συγκρίνουμε την κατάσταση με τα αεροδρόμια, ελάχιστα θίγονται στην Ευρώπη. Δεν θα λοιπόν έχω μία ανάλυση, γιατί είναι αλήθεια ότι ε, στη Βιέννη και στη Φραγκφούρτη, που εγώ δεν θέλω να πηγαίνω εκεί γιατί χάνω τη βαλίτσα μου κατά κανόνα και αν μπορείτε εσείς ε, να προβάλλετε άλλα επιχείρηματα που δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα να τα ξέρω. Όμως εγώ δεν είδα πουθενά να υπάρχει μια αξιολόγηση των κινδύνων και αυτό το βρίσκω απαράδεκτο. Ε, δεν θέλω να φέρω συγκεκριμένα αεροδρόμια, δεν θέλω να το ονοματίσω. Ε, είναι περίπου 7 υπάροχοι στις υπηρεσίες εδάφους σε αυτά τα αεροδρόμια και τελικά συνήθω κάνει κανείς τη βαλίτσα του και για να τη βρει πρέπει να περάσει όλες ώρες ολόκληρες. Brian στο Birmingham, το αεροδρόμιο είναι μια χαρά, έτσι δεν είναι. Αυτό ήταν το ένα. Τώρα πάω στο δεύτερο. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι φάρσα το ότι ξανασυζητάμε το ίδιο θέμα, όλα αυτά που έχουμε ήδη συζητήσει και η συμβαστική πρόταση για λίγα μόνο αεροδρόμιο και να γίνει αυτό ευρωπαϊκός κανονισμός, αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς παραμένουμε στην απόρριψή μας και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με τη μορφή που δίνουμε εμείς την πρόταση, έτσι θα περάσει και στην Ολομέλεια. Ο κύριο ε, Κάλα. Ευχαριστώ και για μένα αυτή η τροποποιημένη πρόταση τη Κομισιόν δεν είναι κάτι που μπορώ να το υποστηρίξω. Και νομίζω ότι και στην επόμενη ψηφοφορία θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα όπω την προηγούμενη φορά. Δεν νομίζω ότι πρόκειται εδώ για καλύτερη νομοθεσία, όπω λέει η Κομισιόν, αλλά περισσότερο για νομοθεσία για να σώσει τα έπιπλα, για να μειώσει τι ζημιέ. Δεν φαίνεται εδώ πέρα να ήταν το απαιτούμενο από την Κομισιόν το να βελτιώσει την κατάσταση, αλλά το να πετύχει μεγαλύτερη φιλελευθερωποίηση της αγοράς. Και ξέρω ότι ακόμα και αν έχουμε τρεις ή τέσσερις παρόχους, μπορούμε να έχουμε καλούς και κακούς παρόχους. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ε, εγγύηση ποιότητας η οποία θα προέλθει από την ποσότητα, μόνο με το να έχουμε περισσότερους παρόχους και η Κομισιόν δεν ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξη για να επιτύχει ποιότητα. Κάτι ακόμα στην περίπτωση που δεν υπάρξει απόρριψη. Η δική μου άποψη, η δική μου θέληση ήταν στα πλαίσια της ε, αναζήτησης ε, συμβιβαστικών λύσεων στην Α2 να υπάρχει και η προσθήκη στο φως των τοπικών συνθήκων αυτό να, να διαγραφεί ώστε να παραμείνουν τα θέματα αυτά στην απόλυτη δικαιοδοσία και διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Αυτό είναι στοιχείο τη επικουρικότητα και εδώ έχετε και ένα σημείωμα τη νομική υπηρεσία για το θέμα αυτό. Επίση, στη συμβαστική τροπολογία σε λατινικό. Αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη αυτοαξυπηρέτηση, οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν αυτοεξυπηρέτηση, θα πρέπει αυτό να θεωρηθεί ότι ήδη είναι μια μορφή φιλελευθεροποίησης και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια διάκριση μεταξύ αυτοεξυπηρέτησης και εξυπηρέτησης από τρίτους. Επομένω, η αυτοεξυπηρέτηση θα πρέπει να είναι τμήμα του δίκτυ, η ύπαρξη τέτοιων εταιριών. Και τρίτον, νομίζω ότι ο ρόλος των ε, αεροδρομίων θα πρέπει να ενισχυθεί για τον συντονισμό των υπηρεσιών εδάφους και επομένως να έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν ανεπαρκή εξυπηρέτηση στο έδαφος και αυτό δεν νομίζω ότι έχει διατύπωθει σωστά. Είναι κάπως υπερβολική αυτή η διατύπωση. Τι θα κάνει λοιπόν, θα πηγαίνει το αεροδρόμιο και θα ρωτάει τους εμπλεκόμενους κατά πόσο λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, επομένως και στην ε, τροπολογία 11 της συμβαστική έχω καταθέσει μια πρόταση για μια απλοποίηση αυτής της διαδικασίας. Αυτά είναι τα σημαντικά σημεία για μένα. Αλλά εγώ πιστεύω αν δεν περάσει η πρώτη τροπολογία, όλα τα άλλα πρέπει να μείνουν στα θέματα της επικουρικότητας. Αλχαντράουι. Θα ήθελα να σας πω αρχικά ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ της καθεστικής τάξης ε, στον τομέα αυτό. Είναι... Δεν είναι ικανοποιητική η νομοθεσία, αλλά δεν μας ικανοποίησε ούτε και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανέκαθεν, ήμασταν υπέρ της ε, ε, αναβάθμισης του κειμένου που αρχικά κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε κάνει κάποια βήματα προόδου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, ε, διότι ανταποκρίθηκε ως επιτοπλίστων στις προσδοκίες μας και η απόδειξη είναι ότι καταλήξαμε σε μια σειρά από συμβαστικέ λύσει. Ο σκιώδη μα, ο κ. Φλέκενστάιν, επίση ε, εξέθεσε τώρα κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε. Επίσης, ε, θα επιθυμούσαμε να επικρατήσει μια μεγαλύτερη ευελιξία ως προς ε, τις επικουρικές ε, υπηρεσίες. Έχουμε καταθέσει και έναν εναλλακτικό κατάλογο ψηφοφοριών. Θα θέλαμε να δίνεται επίσης η ευκαιρία επιλογής ανάμεσα σε δύο παρόχους. Η συμβαστική Α2 ελπίζουμε να εγκριθεί αφορά στην ε, υπεργολαβία η επόμενη θέση που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα θέλαμε να ε, ε, εισαχθεί μέσα στο κείμενο η έννοια της ανωτέρας βίας. Ε, για την ευελιξία που επιθυμούμε, επανέρχομαι ως προς τον αριθμό των παρόχων. Αν γίνει δεκτή η πρόταση που καταθέσαμε, θα μπορέσουμε κι εμείς να υποστηρίξουμε την πρόταση και στην Ολομέλεια η ομάδα μας ομόφωνα θα εγκρίνει την πρόταση. Ελπίζουμε αύριο να υποστηριχθούν αυτές οι συμβαστικές προτάσεις. Σα <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε ότι δεν έχουμε μία ενιαία θέση. Έχουμε μόνο μία ψήφο για το θέμα αυτό από την πλευρά του ΕΛΚ. Έχουμε όμως δείξει την θέλησή μας να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση και όπως είπε ο Σάιντ, ε, συμφωνούμε και εμείς ότι δεν πρέπει να μιλήσουμε μονάχα για τη φιλελευθερωποίηση, αλλά θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από πρόοδο στα κοινωνικά θέματα. Και όποιος εγκρίνει την έκθεση αυτή ως έχει, ψηφίζει κατά των, των πρόοδων στα κοινωνικά θέματα. και για μένα είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν καλύτερες κοινωνικές ε, συνθήκες και να μην παραμείνουμε μονάχα σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό. Δεν σημαίνει το να έχουμε δύο παρόχους στα βελτιώσει τις κοινωνικές συνθήκες. Εγώ δεν νομίζω τώρα ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα για την Κομισιόν αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια, το πακέτο αυτό για τις ε, υπηρεσίες εδάφους, αλλά πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον σε τρει τομεί. και στο μέλλον πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε ένα πιο έντονο διάλογο με τις ε, χώρες μέλη. Για μένα, για να επανέλθω στο θέμα της επικουρικότητας, είναι πάντα η ίστατη λύση. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω ότι είναι αρνητικό, αλλά αν δεν υπάρχει καμιά άλλη δυνατότητα, πρέπει να καταλήξουμε στην ε, επικορικότητα. Αλλά η δική μας δουλειά θα πρέπει να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια καλύτερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να τακτοποιήσουμε τα πράγματα καλύτερα και να μην αφήσουμε να λύνονται όλα στο επίπεδο της επικουρικότητας. Γιατί η επικουρικότητα μας οδηγεί σε 27 διαφορετικές λύσεις στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο καθένας στη χώρα του κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό δεν μπορώ να υποστηρίξω ιδιαίτερα την επικουρικότητα. Δέχομαι τις άλλες απόψεις, αλλά για μένα η ενωσιακή μέθοδος είναι η καλύτερη λύση την οποία ανέφερες και εσύ και δεν πρέπει να καταλήξουμε στο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε προσθέμενη αξία στα κοινωνικά θέματα, στη μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνη και μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια καλή συζήτηση με το Συμβούλιο, γιατί αυτό το πακέτο, όπως έχει αυτή τη στιγμή, έχει πολύ περιθώριο για βελτίωση. Ευχαριστώ. Φώστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και όλους όσους εργάστηκαν σκληρά. Όπως ε, ο Πίτερ Βαντάλεν, θα συμφωνήσω και εγώ για αυτά τα στοιχεία που ανέφερε. Έχουμε όμως ε, και διάφορες ερωτήσεις διευκρινιστικές για τη συμβαστική AIDS τι λέμε ακριβώς που φαίνεται ότι δεν εφαρμόζεται στις περισσότερες επιχειρήσεις και στις περισσότερες βιομηχανίες όπου είναι εμπορικές ή συμβάσεις. Φυσικά θέλουμε να είναι αξιοπρεπείς οι συνθήκες εργασίας, αλλά έχω μία ερώτηση για το άρθρο 12 του κανονισμού. Δέσμευση δηλαδή για την αναδρομική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων. Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό, εάν αποσπαστεί προσωπικό ή μεταφερθεί προσωπικό από τη μία εταιρεία στην άλλη, πώ θα εφαρμοστεί αυτό. Αυτά για το H. Για το J, είναι ένας κανόνας που εφαρμόζεται στους υπεργολάβους και πάλι μιλάμε για τον νομικό εκπρόσωπο για την τηρήση των συλλογικών συμβάσεων. Επίσης θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμβαστική L. Ε, θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι γίνεται με την ανώτερα βία και με τις απεργίες. Ε, όταν ασχοληθήκαμε για την εσωτερική ναυσιπλοεία, μιλήσαμε για τις βασικές εξαιρέσεις και μία από τις βασικότερες για τις αεροπορικές εταιρείε ε, και τα λοιπά είναι ότι η απεργία πάντοτε φαίνεται να εντάσσεται σε αυτή την έννοια της ανωτέρας βίας. Οπότε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η διάταξη Πώ ακριβώ θα εφαρμοστούν οι έκτακτε περιπτώσει ή ανωτέρα βία για να μην γράφονται όλε οι απεργίε ε, σε αυτή τη διάταξη. Γιατί άμα είναι απεργία θα πρέπει να την ονομάζουμε απεργία και αυτό ισχύει για όλου του σχετικού κανονισμού και οδηγίε. Θα ήθελα πρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εισηγητής να μου τα εξηγήσουν αυτά. Ευχαριστώ κύριο Φέρμπερ. Κύριε Πρόεδρε, ελέγχθησαν πάρα πολλά και εγώ θα είμαι σύντομος. Νομίζω πρέπει να προσέξουμε για πρώτη φορά να μην μπερδέψουμε το αίτιο και το αιτιατό. Το αίτιο είναι ότι θέλουμε να ανοίξουμε την αγορά στο αιτιατό, κατά πόσον θα επιτύχουμε κάτι στον κοινωνικό τομέα, νομίζω ότι όλο αυτό είναι οξύμορο. Δηλαδή, ε, δεν θα πετύχουμε τίποτα αν ε, δεν αυξήσουμε τεχνητά τους αριθμούς. Ε, και τίθεται το εξή ερώτημα. Με την κείμενη νομοθεσία, τι πρέπει να αλλάξει. Εξάλλου αυτό ισχύει και για την επικουρικότητα. Δηλαδή, αν πούμε ότι ό,τι απομένει θα ε, ρυθμίζεται επικουρικά με την αρχή της επικουρικότητας. Δεν χρειαζόμαστε νέα οδηγία. Η επικουρικότητα καλή είναι ως ένα μέσο, αλλά για μένα τι το εξή ερώτημα. Γιατί να χρειάζονται όλα αυτά. Έχουμε την νομοθεσία που προσφέρει δυνατότητες. Και θέλω να δείξω και άλλα δύο θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με τους ε, παρόχους. Ε, ένα θέμα που με απασχολεί είναι το εξή υπάροχοι στα διάφορα αεροδρόμια. Γιατί να μπορούν να προβαίνουν ε, σε χρηματοδότηση. Έκανα αυτή την ερώτηση και θα με ενδιέφερε να απαντηθεί. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί στο πλαίσιο ενός μονοπολίου ίσως και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξεκινάει ανταγωνισμός με τιμές ε, και κόμιστρα που όλα αυτά γίνονται εις βάρος των απασχολούμενων και προέρχονται κατ' ουσίαν από το προστατευόμενο μονοπόλιο. Στη Γερμανία, ας πούμε, συμβαίνει αυτό. Το κάνει ένας Ελβετός. Ε, οι Ελβετοί δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο. Και το δεύτερο, όπου έχω κάνει προτάσεις στον εισηγητή, αφορά την ε, διαχείριση των ε, αεροδρομίων. Οι πάροχοι παρεμβαίνουν στις υποδομές. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όλο και περισσότερες εταιρείες εμπλέκονται στην υπόθεση και αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω, με εκπλήσει λιγάκι το γεγονός ότι σε αυτά τα θέματα δεν ψηφίζουμε για μεμονωμένες προτάσεις αλλά για συμβιβασμού. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ τεχνικά τα θέμα. Ε, δηλαδή δεν λέμε καταργείται ο ΑΒΓ πάροχος, αλλά εξετάζουμε ε, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να έχω μία απάντηση, γιατί νομίζω ότι ε, τους τελευταίους μήνες η αντιπαράθεση εμφανίστηκε τελείως διαφορετικά όσον αφορά την επιδότηση και τις ε, χρηματοδοτήσεις ανάμεσα στα διάφορα αεροδρόμια. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα, οφείλεται στην Lufthansa η, η καθυστέρηση στην έλευσή μου. Δεν μπαίνω ούτε καν βαλίτσα, γιατί με βαλίτσα δεν θα ερχόμουν ποτέ. Αλλά εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φέρμπερ για τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μονοπωλίων. Βλέπω ότι η ύπαρξη δύο ή τριών παρόχων θα έχει ένα σαφές αποτέλεσμα. Θα είναι πάντα οι ίδιοι οι οποίοι θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη και εξίσου άσχημα. Και δεν θα υπάρξει αυτό το οποίο υπήρχε προηγουμένως. Και αυτά δεν έχουν καμία σχέση με οι ρυθμίσεις αυτές. Ο επιβάτης ενδιαφέρεται μονάχα για την εξυπηρέτηση, για τις βαλίτσες του, για το και τα κτλ. Αλλά αυτό το οποίο προτείνεται αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό μονοπόλιο. Έχουμε ουσιαστικά και σε αεροπορικές εταιρείε, εκτός από τις συνδέσει μεταξύ των μεγάλων πρωτεύουσων, έχουμε περιφερειακά μονο, μονοπόλια. Αυτό δεν γίνεται. Έχουμε πάρα πολλού μεγάλους σχηματισμούς που έχουν δημιουργηθεί και τα θέματα της ε, διαχείρισης έχουν οδηγήσει σε τεράστιες δομές. Έχουμε λοιπόν τελικά μια οργανωμένη ανευθυνότητα σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών. Επομένως, τελικά αυτό το θέμα δεν έχει επιληθεί με την επεξεργασία και την πρόταση της Κομισιόν. Σας λέω ότι για μένα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα είναι δύο-τρει μεγάλε εταιρείε σε όλη την Ευρώπη, οι οποίε θα έχουν γενική γεωγραφική εξάπλωση και θα μπορούν να παίρνουν λεφτά από ένα αεροδρόμιο και να τα επενδύουν στι υπηρεσίε του σε ένα άλλο αεροδρόμιο. Θα πρέπει να προσέξουμε να δούμε ποιε είναι οι δομέ που δημιουργούμε. Αν Υπάρχει ένα πρόβλημα με ένα από αυτού τους μεγάλους δύο ή τρεις παρόχους, για τρει μέρες θα γίνεται ο χαμός σε όλη την Ευρώπη, αν είναι παρόντες σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα αεροδρόμια. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το, το θέμα, και κάνω μια τελευταία έκκληση, πιστεύω ότι αυτό το θέμα έχει αντιμετωπιστεί με τρόπο που είναι αντιπαραγωγικό, ακόμα και από έποψη νομοθετική. κάνουμε ε, μια ρύθμιση για τα μεγάλα μονάχα αεροδρόμια και τι κάνουμε, από δύο παρόχους πηγαίνουμε σε τρεις παρόχους και αυτό θα αυξήσει περισσότερο το δυνητικό χάος. Δεν είναι καλή νομοθεσία αυτή, δεν είναι καλή διαδικασία νομοθεσίας. Λοιπόν, ας την αφήσουμε κατά μέρο όλη αυτή τη ρύθμιση. Θα πρέπει αντίθετα να δώσουμε περισσότερη έμφαση <clears throat> στο να μην υποσκαφθούν περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων στα αεροδρόμια και δεν θέλουμε να ανοίξουμε πόρτες οι οποίες δεν φέρνουν την παραμικρή βελτίωση. Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους ε, εργαζόμενους και όχι να τη χειροτερέψουμε. Λοιπόν, ας μην το ε, προχωρήσουμε περισσότερο αυτό το θέμα. Κύριε Φίγκελστάιν, είπατε ότι θέλετε και πάλι να λάβετε το λόγο, αλλά μπορείτε να είστε σύντομο, είπατε. Μπορώ. Γιατί έχει περισσότερο νόημα από το να διαβάζω μακροσκελείς λόγους οι οποίοι απευθύνονται στους συναδέλφους που δεν μ' ακούνε. Εγώ ε, θα ήθελα να σταθώ σε αυτά τα οποία ελέγχθηκαν προηγουμένως. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Και υπάρχει πάντα δυνατότητα οι σκιώδεις εισηγητές να μπορέσουν να συζητήσουν και πάλι και αν ε, συμφωνεί και ο κύριος ε, Ζασάντα μπορούμε να το κάνουμε και απόψε ακόμα. Δεύτερον, για την κατεύθυνση που αναφέρει η κυρία Λίχτεμπεργκ. Η βελτίωση των κοινωνικών στάνταρ. Η βελτίωση των προτύπων ποιότητος. Αυτό είναι το μόνο εγχείρημα το οποίο κατά την άποψή μου έχει νόημα να μας απασχολήσει. Και συμφώνω με αυτά. Τώρα, το να επιβάλλουμε μία περιττή υποχρεωτική επέκταση της φιλελευθερωποίησης, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εγώ μπορώ να δεχτώ. Και δεν μπορεί αυτό να είναι το αντίτιμο για οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση. Και ένα τελικό ερώτημα. Για τον κύριο Γκρός. Είπατε ότι χαίρεστε με, για την ευκαιρία να συζητήσουμε με το Συμβούλιο, γιατί λέτε ότι μπορεί να προκύψει κάποια βελτίωση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε ποιο τομέα και σε ποιο βαθμό μπορείτε να περιμένετε κάτι από το Συμβούλιο για αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις. Μα όλοι θέλουν να ξαναδευτερολογήσουν. Κύριε Μάισνερ. Το πρόβλημα με κάθε ερώτημα είναι ότι απαιτεί μια απάντηση και δεν τελειώνει ποτέ η συζήτηση. Η κυρία Μάισνε πρώτα, παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Δεν θα έχουμε δευτερολογίε μόνο για διευκρινήσει θα σα δίνω το λόγο. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα είμαι σύντομη, γιατί ε, μοιάζει να μην υπάρχει καμία βελτίωση. Αυτό ε, που έχει σημασία είναι ότι το θέμα δεν είναι ο αριθμός των παρόχων, αλλά ε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να τα βελτιώσουμε, όπως ε, την ποιότητα των προδιαγραφών ή ε, τις υπεργολαβίες. Αυτά δεν ρυθμίζονται καλά. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν προς όφελος των επιβατών. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει τον κόπο τους ε, συμβιβασμού που μας προτείνει η συγητής να τους δούμε πολύ προσεκτικά και ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε αύριο. Ε, Κοιτάξτε, συνάδελφε Φλέκενστάιν, εσείς δηλαδή τι θα κάνετε αν απορριφθούν οι συμβαστικές προτάσεις. Ε, θα καταψηφίσετε. Ναι, στην τελική θα καταψηφίσω. Εσείς προσωπικά ή η πολιτική σας ομάδα. Ε, προφανώς δεν με ενδιαφέρει η προσωπική σας ψήφος, της πολιτικής σας ομάδας με ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, ό,τι και να ρωτήσετε μου είναι παντελώς αδιάφορο. Στη δική μου την επιτροπή οι γίνονται μέσω του Πρόεδρου, όχι απευθείας. Εάν λοιπόν θέλετε να πείτε κάτι θα ζητήσετε ε, το λόγο από τον Πρόεδρο και όχι διάλογος ε, με τον κύριο Φλέκενστάιν ε, απευθείας. Ο κύριος Μπόλντουιν, εκ μέρους της Κομισιόν, παρακαλώ. Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί έχω μιλήσει εδώ πολλά και στην Επιτροπή σας και είναι γνωστέ οι απόψει μας για όλα αυτά τα σημεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές βοηθούς που εργάστηκαν στην, στα σιβηρικά ορυχεία των υπηρεσιών εδάφου και έχουν χύσει αίμα. Λοιπόν, απαντώ σε ερωτήσει. του κ. Βαντάλεν. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο όντω έχει καταλήξει σε μια γενική προσέγγιση για τι υπηρεσίε εδάφου. Υποστηρίζει την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέποντα τι εφαρμοστέ συλλογικέ συμβάσει και την διαδικασία διαγωνισμών. Ευχαριστούμε, κύριο Σασάρα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πάλι κοιταζόμαστε όλοι μέσα στην αίθουσα ε, χωρίς να καταλαβαίνόμαστε. Ε, το έγγραφο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά τελικά όλες οι συζητήσεις περιστρέφονται ε, γύρω από τον αριθμό των παρόχων. Έχω διαβάσει εκατοντάδες φορές το έγγραφο και πιστέψτε με δεν είναι αυτό το σημείο κλειδί και γι' αυτό πρότεινα δύο εναλλακτικές εκδοχές της συμβαστικής Α. Μία εκδοχή που αποφασίζει το κράτος μέλος, αν θέλει να διευρύνει την αγορά και τη δεύτερη εναλλακτική, όπου περιορίζουμε στους τρεις ε, τους ε, παρόχους ε, για κάποιους αερολιμένες μέχρι τα 15 εκατομμύρια. Ξέρετε, στη χώρα μου έχουμε 40 εκατομμύρια και δεν υπάρχει αερολιμένες όπου υπερβαίνουμε τα 15 εκατομμύρια επιβατών ως προς την κίνηση των αεροδρομίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο υψηλό είναι το ανώτατο όριο. Ισχύει για τους μεγαλύτερους αερολιμένες όταν κάποιος μιλάει για άκρατη απελευθέρωση τη αγοράς, νομίζω ότι πραγματικά δεν έχει διαβάσει την έκθεση. Ε, ας ε, απευθυνθώ συγκεκριμένα στους συναδέλφους από την ΚΟΕ ή από τους Πράσινους. Ε, μας μιλάνε για κάποιες διατάξεις προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων ε, που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τους προσφέρουμε κάτι που δεν υπάρχει προς το παρόν ε, στα κράτη-μέλη. Ε, και όταν μας εκβιάζουν με τους δύο ή τρεις παρόχους ε, και ότι θα καταψηφίσουν ολόκληρο το έγγραφο μόνο και μόνο για το θέμα του αριθμού των παρόχων, δεν καταλαβαίνω ακριβώς ε, τη θέση τους. Αν κάποιος έχει διαβάσει έστω και μία φορά την έκθεση θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα και αν θέλουμε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες οφείλουμε να εγκρίνουμε αυτό το έγγραφο δίχως αυτό κανένα αεροδρόμιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφ' δεν θα υποχρεώνει τους παρόχους να παράσχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Δεν θα προβλέπονται οικονομικές κυρώσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης και καταλαβαίνουμε φαίνεται ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση στα αεροδρόμια. Μέσα από αυτό το έγγραφο παρέχονται όλες οι προϋποθέσεις ε, για να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες ε, και απευθύνομαι σε αυτούς που θέλουν να αναπέμψουν ε, το έγγραφο στην Επιτροπή. Μιλάτε για τον αριθμό των παρόχων και ξεχνάτε και τα κοινωνικά δικαιώματα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτή την, με αυτό το έγγραφο λέμε ότι μέσουσες της κρίσης χρειαζόμαστε περισσότερες θέσεις απασχόλησης, καλύτερες θέσεις απασχόλησης προτείνουμε 27 διαφορετικές διαδικασίες διαγωνισμών και έγκρισης για την αδειοδότηση. Με αυτό το έγγραφο όλα αυτά αλλάζουν άρδιν και με την εφαρμογή του εγγράφου ε, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να καταψηφίσει αυτό το έγγραφο. Ίσως το πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάω γερμανικά, γιατί από ό,τι φαίνεται η διαχωριστική γραμμή, ε, η κόκκινη γραμμή είναι τα γερμανικά. Θα ήθελα λοιπόν να βελτιωθεί η κατάσταση χάρη σε αυτό το έγγραφο, γιατί δεν είναι καθόλου ικανοποιητική σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν μετά τη σημερινή συζήτηση να έρθουν όλοι οι σκιώδεις, ε, θα σας, ε, να τους κεράσω ένα καφέ για να συνεχίσουμε να συζητούμε τις συμβαστικές ε, λύσεις. Εδώ και ένα χρόνο τη συζητάμε, θα ήθελα να το υπενθυμίσω εν παρόδο και τώρα ε, πέντε λεπτά πριν το τέλος ε, λένε κάποιοι ότι μπορούμε και να το βελτιώσουμε. Αν μπορούμε, ελάτε για καφέ και θα τα βρούμε. Ο κύριος Σίμψον, μπορείτε σε αυτά τα λεπτά να πιείτε πολλούς καφέδες μέχρι να τα βρείτε για τις συμβαστικές. Μάλιστα... Αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής να θυμηθούν να φέρουν τις κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν θα επιτρέψω ε, ανάταση χειρός για τις ηλεκτρονικές ε, ψηφοφορίες ε, γιατί ορισμένε φορές ε, η διαφορά είναι λίγες ψήφοι. Δεν θα το επιτρέψω λοιπόν. Σας το υπενθυμίζω να έχετε φέρει τις κάρτες σας και θα ζητήσω από την Γραμματεία να το υπενθυμίσει και στους συναδέλφους που απουσιάζουν σήμερα. Επόμενο σημείο είναι προϋπολογισμός 2014. Η κυρία Γένσεν είναι η γενική εισηγήτριά μας, δεν είναι εδώ, οπότε διακόπτουμε μέχρι ότου να καταφτάσει στις 4 η ώρα για, το, για τη γενική συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2014.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

Okay, colleagues. Πάμε συνάδελφοι. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η παρουσίαση της Γενικής Εισήγησης για τον προϋπολογισμό του 2014, η Άννη Γιένσεν, όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά. και είμαστε σε αυτή την τόσο παράξενη αίθουσα. Δύσκολα βλέπω χωρίς τα κιάλια μου τους ε, άλλους βουλευτές, αλλά ευχαριστούμε πολύ, Αν, για την παρουσία σου εδώ σήμερα το απόγευμα. Ξέρω ότι πέρσι είχαμε μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Λαβία και την προηγούμενη εβδομάδα επίσης στην Ολομέλεια έλαβε χώρα μια συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η κυρία Αιάλα Σέντα και ο κύριος Ρίπλεϊ θα ξεκινήσουν και την συζήτηση, τον τριγωνικό διάλογο για το σχέδιο Connecting Europe. Επομένως, οι σχέσεις μας με την Επιτροπή Προϋπολογισμών συσφίγγονται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε για να αποκομίσουμε τους απαραίτητους για μας πόρους. Δεν πειράζει όμως, αν μπορείτε να μας δώσετε τις απόψεις σας, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Μπράιν. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στην αγαπημένη μου επιτροπή, παρότι ε, αποχώρησα. Είναι ιδιάζουσα η κατάσταση με τον προπολογισμό αληθεύει αυτό. Δεν έχουμε το πολιετές νομικό πλαίσιο, δεν έχουμε τη σχετική νομοθεσία και άρα υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά. Μπορώ όμω να πω ότι είναι σε καλά χέρια η Επιτροπή Μεταφορών λόγω των δικών σου δεξιοτήτων, Μπράιαν, και των ικανοτήτων των σκιωδών των δύο μεγάλων ε, πολιτικών ομάδων. Είμαστε πλέον ε, πολύ άριθμοι ε, εμείς που κατανοούμε τις προτεραιότητες από πλευράς μεταφορών. Ένα βασικό ζήτημα είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe και σίγουρα στα πλαίσια των συζητήσεων για το νομικό πλαίσιο είναι το καταλητικό ζήτημα που θα ορίσει όχι μόνο το τελικό ποσό αλλά και την κατανομή στις τρεις, στους τρεις επιμέρους τομείς. Θα μας απασχολήσει λοιπόν και στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να είμαστε όλοι σε στενή ε, επαφή αλλά και για τον ετήσιο προϋπολογισμό θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να το αναδείξουμε σε προτεραιότητα. Άλλο σημαντικό σημείο, οι οργανισμοί. Ε, πολύ συχνά ε, το Συμβούλιο καταλήγει σε πολύ περίεργες ε, αποφάσεις με οριζόντιες ε, περικοπές, δίχως να επισέρχεται σε μία ε, ενδελεχέστερη μελέτη των αναγκών του κάθε οργανισμού. Και αυτό θα μας απασχολήσει λοιπόν. Αύριο θα γίνει ο πρώτος τριμερής διάλογος Κοινοβουλίου Συμβουλίου Επιτροπής για τον ε, προϋπολογισμό του 2014 θα συζητήσουμε και τη μεθοδολογία εργασίας ε, μεταξύ άλλων. Έχει, έχω την εντύπωση ότι το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει, δεν έχει συνειδητοποιήσει τις νέες αρμοδιότητες συνθήκης της Λισαβόνας, γιατί το πνεύμα της επιτάσσει ότι έχουν ίσα δικαιώματα τα δύο θεσμικά όργανα ε, κατά τη διαστολή με το παρελθόν ε, που είχαμε στον τελευταίο λόγο για όλα τα υπόλοιπα εκτός από τη Γεωργία. Ίσα δικαιώματα λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει μία σειρά συζητήσεων για κάθε επιμέρους γραμμή του προϋπολογισμού ουσιαστικά. Τι συμβαίνει όμως. Το Συμβούλιο δεν φαίνεται να είναι έτοιμο να συζητήσει ή να διαπραγματευτεί μαζί μας την 21η μέρα, δηλαδή αυτή η περίοδος των 21 ημερών μετά την έγκριση της θέσης μας και θα ε, μιλάμε για τις πληρωμές και στη συνέχεια μας λένε ναι, αποφασίζουμε το γενικό ποσό και εσείς αποφασίστε για την κατανομή. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και δύο από τις τρεις φορές αυτό συνέβη γιατί λίγο κόντεψαμε να μην έχουμε καν εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τελευταία στιγμή συμβαίνουν όλα χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος. Νομίζω μας χρειάζεται μια καλύτερη μεθοδολογία εργασίας, ούτως ώστε σε, ε, ε, νωρίτερα και όχι την τελευταία στιγμή να εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια. Λοιπόν, ζητώ την υποστήριξή σας, όπως και όλων των υπολείπων επιτροπών, για να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να γνωρίζουμε ποιε είναι οι λεπτομέρειες κάθε ζητήματος για να προβάλλουμε τις δικές μας προτεραιότητες. Πάντως, ε, όλα όσα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών είναι ζητήματα που πραγματικά θα μας απασχολήσουν και θα είναι ιδιαίτερα ε, επίμαχα για τον προϋπολογισμό του 2014. Brian Simpson, ευχαριστούμε. Αν ε, η κυρία Ντυράν είναι η συγγήτριά μας για τον προϋπολογισμό, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε αγαπητή Άννα για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Ξέρουμε λοιπόν ότι είναι ιδιάζουσα η κατάσταση όπως προανέφερες. Θα επεξεργαστούμε το χρονοδιάγραμμα για το προϋπολογισμό του 2014. Ταυτόχρονα όμως είναι ομιχλώδες το τοπίο για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και αν θα εγκριθεί το ε, πολιετές αυτό πλαίσιο, δεν ξέρουμε πότε, μέχρι το τέλος του 2013, αν θα υπάρξει συμφωνία και ποια θα είναι αυτή η συμφωνία. Και καλό θα ήταν να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην καταλήξουμε συμφωνία στο Κοινοβούλιο και τότε θα χρησιμοποιήσουμε τα τα όρια του 2013 και όχι τον προπολογισμό το 2014. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η δική σου άποψη προτού εισέλθουμε στο περιεχόμενο και στις λεπτομέρειες των θεματικών ενωτήτων, κάτι που θα συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή, πώς κατά τη γνώμη σου συνδέεται ο, αυτός καθ' αυτός ο προϋπολογισμός το 2014, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ε, το, η άλλη πτυχή, το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας ε, την Ευρώπη, είναι λοιπόν η διάσωση περίπτωση μόνο και μόνο προς το χρονοδιάστημα Πώ ε, Πώς ακριβώς ε, εργαζόμαστε πρέπει να μας απασχολήσει πρώτα η μεθοδολογία και στη συνέχεια το περιεχόμενο, δηλαδή ποιε προτεραιότητε θα προτάξουμε εμείς ως Επιτροπή Μεταφορών για τον προπολογισμό του 2014. Πρέν Σίμψον, ευχαριστούμε ο κύριος Ντερίκη Ελκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τα ήδη λεχθέντα. Είναι σαφές όμως ότι το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι επί τη βάση ποιου εγγράφου η συγγήτρια η αν θα μπορέσει να φέρει σε πέρα στο έργο της. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε επί ποια βάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση προπολογισμού για το 2014. Είναι υποχρεωμένη να το κάνει γιατί δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για τι πολιετές δημοσιονομικές προοπτικές. Και επομένως η Κομισιόν θα πρέπει να καταθέσει μια πρόταση επί τη βάση τη δική τη πρόταση για το, δικό, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Άσκηση σουρεαλισμού λιγάκι. Ξέρουμε ότι μέχρι τότε μπορεί να υπάρξει κάποια τροποποίηση και συμφωνία με το Συμβούλιο και μπορούμε να καταλήξουμε επίσης να μεταφέρουμε απλώ τα στοιχεία του 2013. Αλλά το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα προτείνει η Κομισιόν ε, ώστε να είναι το αρχικό σημείο κίνησης για την εισηγητριά μας. Δεν ξέρουμε λοιπόν προς τα που αρμενίζουμε σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Όποια και να είναι με πάση περιπτώσει αυτή η βάση η οποία θα προταθεί, όποια και να είναι τα προβλήματα τα οποία τίθενται για μας, μας ενδιαφέρει το θέμα, το θέμα της ε, χρηματοδότησης των επενδύσεων του Connecting ε, Europe Facility, το Συμβούλιο έχει περικόψει κατά 40% αυτό τον προπολογισμό που μου φάνηκε ότι είναι υπερβολικό και νομίζω ότι αν υπάρχει μια τόσο μεγάλη ε, μείωση, απομείωση των κονδυλίων, αυτό οδηγεί κατά ανάγκη σε αλλαγή της νομικής βάσης. Δεν μπορούμε να πετύχουμε τα ίδια με προπολογισμό ο οποίος είναι τόσο πολύ ψαλιδισμένος. Ίσως πρέπει να ρωτήσουμε το Συμβούλιο ποια είναι τα, ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες αυτής της περικοπής, εάν το Συμβούλιο λοιπόν έχει να, έχει να κάνει κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το Connecting Europe Facility για τα θέματα μεταφορών. Υπάρχει το γενικό θέμα των πληρωμών το οποίο δεν έχει επιληθεί και το οποίο μας ε, επιβάλλεται με ένα πολύ σκληρό τρόπο στον προϋπολογισμό του 2014. Θα έχουμε μάλλον 16 δισεκατομμύρια τα οποία δεν θα έχουν ε, επιληθεί σε σχέση με τη δυνατότητα πραγματικής του εκταμείευσης. Δεύτερον, υπάρχει μια ομάδα θεμάτων μέσα στα πλαίσια και των δημοσιονομικών προοπτικών και του ετήσιου προϋπολογισμού του 2014 που θέτει προβλήματα. Για το δικό μας προϋπολογισμό, όπως είπε και η Άν, το θέμα των αποκεντρωμένων φορέων παραμένει ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ο προϋπολογισμός μας να είναι μικρότερος από τον πετσινό τη στιγμή που έχουμε αυξήσει τις αρμοδιότητες και το έργο των αποκεντρωμένων φορέων και στο τέταρτο πακέτο έχουμε προτάσεις για τον Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Φορέα που πρέπει να προωθηθούν αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε <clears throat> ανάλογα τα, τη χρηματοδότηση αυτού του φορέα. Επομένω, για αυτό το φορέα, όπω και για άλλου, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του όταν έχουμε μείωση του προπολογισμού. Και ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό μα ε, αφορά ιδιαίτερα, είναι ο ορίζον 2020. Ξέρουμε ότι ο προπολογισμό των μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι μεταφορέ και για τα θέματα μεταφορών. Η πρόοδο ιδίω στο συνδρομικό κομμάτι, είδαμε ότι ο προπολογισμό ή μάλλον η πρόταση προϋπολογισμού για τον ορίζοντα 2020 έχει μειωθεί, έχει μειωθεί με συγκεκριμένες ενέργειες για τα θέματα μεταφορών τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Και έχουμε και γενικού χαρακτήρα δυσκολίες στον ετήσιο προπολογισμό που έρχονται σε αντίφαση με τις εξαγγελτήσεις γενικές ε, πολιτικές όπως είναι η επίτευξη στόχων για το περιβάλλον. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι οι οποίοι παραμένουν μέσα στο κείμενο της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ και είναι αντικείμενο γενικής συμφωνίας μεταξύ μας όταν μειώνεται ο προπολογισμό παράλληλα. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημείο αναφοράς για τον προϋπολογισμό, αυτό είναι γενικό θέμα, και ξαναθέτω το ερώτημα προς την Κομισιόν. Επί ποιας βάσης θα προτείνει ένα προσχέδιο προϋπολογισμού η Κομισιόν, τώρα πρέπει να το ξέρουμε αυτό, για το 2014. Και η δεύτερη πρόταση, δεύτερο ερώτημα είναι μάλλον, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα με πολύ λιγότερα χρήματα. Και εδώ θα πρέπει το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του και να πει σε ποιους τομείς θα πρέπει να ε, παρετηθεί μιας ομάδος στόχων. Θα πρέπει το Συμβούλιο να καταλάβει και να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές του αντιφάσεις. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν προς το παρόν. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γκάντε Ζεντόπια, για το S&D. Ευχαριστώ. Μπορώ να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Ρίκια. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Και όπως ε, είπαν και οι άλλοι συνάδελφοί μου και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, γιατί φαίνεται ότι εδώ <clears throat> έχουμε βρεθεί όλοι μαζί για να μιλήσουμε για τα θέματα των προϋπολογισμών μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε για τις προτεραιότητες του 2014 όταν δεν έχουμε καν το δημοσιονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να εγγραφεί αυτή η επιλογή προτεραιοτήτων. Αν υπάρξει τελικά μια πρόταση για την ε, θέση του Συμβουλίου ή δεν υπάρχει συμφωνία και πρέπει να συνεχίσουμε για το 2014 το προηγούμενο πλαίσιο, η διαφορά θα είναι 10 δισεκατομμύρια. Τόσο μεγάλη διαφορά δεν υπάρχει στη γεωργία ή στα διαφορετικά ταμεία, αλλά υπάρχουν σε πάρα πολλού τομεί που ενδιαφέρουν τη δική μα επιτροπή, όπω είναι το Connecting Europe Facility ή Horizon 2020, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την επιτροπή μα. Έτσι είναι πάρα πολύ πολύπλοκα τα πράγματα. Μπορεί να είναι σαφεί για μα οι προτεραιότητέ μα, είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε την τελική κατανομή των κονδυλίων που θα αποφασιστούν. Το λέμε αυτό κάθε φορά στο Συμβούλιο. Δεν μπορούν να γίνονται γραμμικέ περικοπέ γιατί πάντα υπάρχουν προτεραιότητες και ανάλογα με τα πόσα χρήματα έχουμε, προτιμάμε να τις κατανείμουμε με τον α ή με τον άλλο τρόπο. Αν έχουμε λοιπόν στο Connecting Euro Facility περικοπές 21 δισεκατομμύρια, εδώ πρέπει να ξανασκεφτούμε από την αρχή την κατανομή των κονδυλίων αυτών. Σε ό,τι αφορά το συνολικό ποσό, το Κοινοβούλιο ήδη εξέφρασε την άποψή του την εποχή της έκθεσης Σούρε αλλά κάποτε θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το συνολικό ποσό και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συμφωνία το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να κατανείμουμε αυτές τις περικοπές. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με γραμμικό τρόπο, θα πρέπει να μας πει η Κομισιόν πού βρίσκεται η προτεραιότητά της, αν θέλει να δώσει περισσότερα στην ενέργεια, στις μεταφορές ή στις τηλεπικοινωνίες, στο Connecting Euro Facility, παραδείγματος χάρη. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα θα παίξουν μεγάλο ρόλο στην απόφασή μας. Και υπάρχει επίσης και το πρόβλημα των πληρωμών. Εδώ και τρία χρόνια σούρνουμε αυτά τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ ελλείμματος από τα προηγούμενα χρόνια και δεν ξέρουμε πώς θα επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Ούτε φέτος ούτε του χρόνου θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό γιατί δεν βλέπουμε το Συμβούλιο να αλλάζει η αντιμετώπιση όπως έλεγε και η κυρία Γέννησε στην αρχή. Τελικά μετά από ένα χρόνο που εργαζόμαστε για προτεραιότητες και έγγραφα και το ένα και όλα αυτά Όλα αυτά στο τέλος συνοψίζονται σε ένα ποσό το οποίο είναι η κόκκινη γραμμή για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καταφέρνει να τους αλλάξει μυαλά. Εμείς τελικά καταλήξαμε το 2012 να έχουμε 16 δισεκατομμύρια έλλειμμα και δεν πιστεύω ότι αύριο στο τριγωνικό διάλογο θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα, τουλάχιστον να μπορέσουμε να θέσουμε κάποιε βάσει εργασία για τι μελλοντικέ συνεδριάσει και να συμφωνήσουμε γιατί θα εργαστούμε, γιατί αν έχουμε πάρα πολλέ προτεραιότητε, τελικά αυτό δεν σημαίνει περισσότερα χρήματα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να εφαρμοστούν τα προγράμματα ή όχι. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης, τότε δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. πρόσφατα στην Ολομέλεια, όταν συζητούσαμε για τις γενικές κατευθύνσεις, η πιο συνηθισμένη λέξη που αναφέρθηκε από όλου ήταν η αβεβαιότητα, γιατί δεν ξέραμε πάνω σε ποια αριθμητικά στοιχεία εργαζόμαστε και ξέρουμε ότι αυτά τα στοιχεία μπορεί να επικύρουν στην πραγματικότητα πάρα πολύ. Συζητάμε λοιπόν στον αέρα και μόνο όταν υπάρξει κάποια συμφωνία με το Συμβούλιο θα ξέρουμε με τι αριθμητικά ποσά πραγματικά παίζουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που την έκθεση αυτή θα την κάνει η κυρία Γένσεν, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα των μεταφορών ε, και βεβαίως ε, φέτος ε, δεν μπορεί κανείς να χαίρεται που θα είναι εισηγητής ε, για τον ε, προπολογισμό, διότι ακόμα δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει με το πολιτέ σε δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο το απέρριψε το Κοινοβουλίο και πολύ σωστά νομίζω, γιατί αναφέρθηκε ότι οι περικοπές που έγιναν από το Συμβούλιο είναι απαράδεκτες και επίσης ε, Θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία για να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό. Και βεβαίως πρόκειται για τα έτη 14 έως 20, άρα δηλαδή πρόκειται ήδη για του χρόνου. Όσον αφορά το Connecting Europe Facility, εκεί ε, μας έκοψαν μόνο το 1 τρίτο, καλά τα πήγαμε. Ε, στην ψηφιακή ατζέντα ε, περικόπηκαν τα 8 ένατα, που είναι πολύ χειρότερα. Το Connecting Europe Facility είναι μια πρόταση που συνδυάζεται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών με τα TNT. Όσον αφορά τώρα λοιπόν τις ε, μεταφορές, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδιαίτερη προοπτική για το μέλλον και ο, ο, κύριος Ρικέ έθιξε το Horizon 2020 και εκεί πρόκειται για κάποιες αναλλακτικέ λύσεις του μέλλοντος που όμως μας τις αφαίρεσαν για να μην αναφερθώ καν στους ε, διάφορους οργανισμούς με μεγάλη ανυπομονησία να δω τι θα γίνει τόσο όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο όσο και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ε, να βολιδοσκοπήσουμε, να δούμε λιγάκι τι μπορεί να γίνει και βεβαίως όσον αφορά εμάς τις μεταφορές. Ευχαριστώ την Επιτροπή Προπολογισμών, όλους όσοι εργάζονται στην Επιτροπή αυτή και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε το δικό μας μάτι και το δικό μας αυτή στην Επιτροπή αυτή. Ο κύριος Ζήλερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με τους υπολείπους. Ε, δεδομένης εμπειρίας της Αν Γένσεν στην Επιτροπή Μεταφορών και στον προϋπολογισμό είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που έχει αναλάβει ε, ως εισηγήτρια για τον ε, προϋπολογισμό. Έχω την εντύπωση ότι η απόφαση και το ψήφισμα του, της περασμένης εβδομάδας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, εκφράζει τις αντιρρήσεις ε, του Κοινοβουλίου για τα μέτρα ευελιξίας σε αυτό τον προϋπολογισμό. Θεωρώ λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση που είχε κάνει για τον προϋπολογισμό το 2014 θα έπρεπε λογικά να αναθεωρήσει ε, τα σχέδιά της στον τομέα των μεταφορών. Ε, Φερρυπίν, ε, χρειάζεται προσαρμογή διότι δεν έχουμε επαρκή κονδύλια για να τα υλοποιήσουμε συμπεριλαμβανομένου και του χρηματοδοτικού μέσου συνδέοντας την Ευρώπη. Το Συμβούλιο με σαφήνεια έχει τοποθετηθεί για τους πόρους που θα χρησιμοποιήσουμε για τη χρηματοδότηση για όλα τα επιμέρους σημεία. Λοιπόν, δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε να γίνουν προσαρμογές στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι συγκητές θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να το επιτύχουν. Ε, θα πρέπει επίσης ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει πάρα πολλά προγράμματα ε, στο Connecting Europe. Έχουμε αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των προγραμμάτων σε σχέση με την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι ρεαλιστικές οι προσδοκίες μας για το 2014. Είναι ανέφικτο ε, χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα. Ενδεχομένω θα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε τον κατάλογο όλων αυτών των προγραμμάτων ή αλλιώ ε, να αφήσουμε στα κράτη-μέλη τη διακριτική ευχαίρεια, αν το επιθυμούν, να συγχρηματοδοτούν κάποια από αυτά τα προγράμματα. χρησιμοποιώντας ε, εθνικά κονδύλια. Ίσως αυτό δεν ισχύει για το Connecting Europe, αλλά και το ίδιο το Συμβούλιο ε, ε, δεν ε, είναι μάλλον υπέρ αυτής της άποψης. Για τους οργανισμούς, στα πλαίσια του τέταρτου πακέτου, όπως είπε ο Επίτροπος Κάλλας, οι ίδιες οι σιδηροδρομικές ε, μεταφορές ε, αρκετά επικερδίσουν, ώστε εν μέρει να χρηματοδοτηθεί ο αρμόδιος ε, οργανισμός. Ίσως θα έπρεπε να επιδιώξουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους ε, που θα πορεύει από τις δραστηριότητες ε, των οργανισμών, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο τμήμα ε, του προϋπολογισμού τους. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριο Γκρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Αν για όλα αυτά τα οποία είπε. Ο προϋπολογισμός είναι στα πολύ καλύτερα χέρια που μπορεί να βρεθεί με την ε, ΑΝ. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλά να κάνουμε για να πείσουμε το Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Εγώ πιστεύω ότι εφόσον θα πρέπει να κάνουμε σαφές ότι δεν συμφωνούμε με τη θέση του Συμβουλίου. Επομένως, εμείς δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε περικοπές στον εαυτό μας αλλά και αυτό που είπε η Άιντεν προς την Κομισιόν είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζω ότι η Κομισιόν δεν θα ξεκινήσει από την απόφαση του Συμβουλίου ως ε, θέση κίνηση, αλλά από τη δική της πρόταση για τον προπολογισμό του 2014. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Ρικέρ, που είναι οι, οι πιστώσεις πληρωμών. Δεν μπορεί τώρα μια επιχείρηση να μην ξέρει αν θα πληρώσει του χρόνου είσαι υποχρεώσει ή όχι. Αυτό ισχύει για όλε τι επιχειρήσει. Δεν μπορεί λοιπόν μια επιχείρηση να λειτουργεί χωρί να ξέρει αν θα μπορέσει να πληρώσει. Εμεί σωρεύουμε τώρα χρέη και καθυστερήσει πληρωμών. Αυτά τα 16 δισεκατομμύρια όπω ελέγχθη στον τομέα μα αυτό. Και πρέπει κάποιο να αναλάβει την ευθύνη σε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρξει κάποια. Ε, κάποια λύση για αυτά. Και δεν μπορούμε όταν βάζουμε πιστώσει πληρωμών στον προπολογισμό αφορούν τα προηγούμενα ποσά που έπρεπε να πληρωθούν ή αφορούν νέα σχέδια. Χρειάζεται λοιπόν να πάρουμε κάποιους ψυχιάτρους για να βοηθήσουν τους πολιτικούς στην Ευρώπη, γιατί έχουν έρθει τα κράτη-μέλη, έχουν κάνει προτάσεις για το Connecting Europe, έχουν θέσει προτεραιότητες, συμφωνούν μαζί μας για το γεγονός ότι θα ήταν πολύ καλύτερα να έχουμε μια καλύτερη υποδομή συνδεδομικών ε, γραμμών, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλουν να μας δώσουν τα κονδύλια για όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουμε εδώ πέρα μια σχιζοφρενική αντίφαση. Όλα αυτά τα οποία περιμένουμε από τη μια μεριά από την Ευρώπη και όλα αυτά από την άλλη μεριά που δεν δίνουμε κονδύλια για κάτι τέτοιο. Εμείς δίνουμε λοιπόν 1% για να καλύψουμε αυτά τα οποία δεν γίνονται με τα άλλα 99% από το ΑΕΠ της Ευρώπης. Πρέπει επομένως να παραμείνουμε σε αυτά τα οποία έχουν προταθεί από την Κομισιόν και όχι από τον πετσοκομμένο προπολογισμό του Συμβουλίου και δεν μπορούμε να αλλάξουμε από τη μια μέρα στην άλλη τον προϋπολογισμό κατά 20% χωρίς να καταστρέψουμε σημαντικά σχέδια. Και γι' αυτό λέω ότι χαίρομαι για τη συζήτηση με το Συμβούλιο, όπου το κάθε κράτος θα πρέπει να αποδεχθεί την διαγραφή σχεδίων που του είναι προσφυλή. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πιο ρεαλιστική συζήτηση. Κράμερ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια για το ότι επανήλθε η Αν στην Επιτροπή Μεταφορών. Προφανώς και παρακολουθούσε πολύ καλά τα θέματα, αλλά τώρα χαιρόμαστε πολύ ε, που είναι κοντά μας. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπε. Κοιτάξτε, είναι παντελώς αδιάφορο το πόσα χρήματα θα πάρουμε, πόσα θα περικόψουν, πόσα θα προσθεθούν. Ένα πράγμα είναι σαφές. Ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Κομισιόν, αλλά ούτε και το Κοινοβούλιο δεν θα ε, παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα και να διερωτώνται ε, κατά πόσον μπορεί να χρηματοδοτηθεί ή όχι. Κοιτάξτε, ε, υπάρχουν όπως ξέρετε πέντε δις και υπάρχουν ε, υπάρχει μια σειρά προγραμμάτων. Αυτό συμβαίνει στη Γερμανία και το συμβαίνει και στην Ευρώπη. Και θα πάρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Στην τελευταία περίοδο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν ήθελαν 20 δι για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Πήραμε 8, περίπου τον τρίτον. Και διαγράφηκε μήπως ένα project, ούτε ένα, τίποτα πάμε στο Connecting Europe Facility. Εδώ διαγράφηκε μόνο το 1 τρίτο. Δεν χρειαζόταν όμως ε, να διαγραφεί τίποτα και τελικά στην πράξη δεν έγινε τίποτα και πολλοί ζητάνε και άλλα προγράμματα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Ε, θα σας πω κάτι που μπορείτε να διαγράψετε. Πρόκειται για τη Στουτγάρντι, όχι όμως για τον περίφημο σταθμό. Πρόκειται για μια διαδρομή Στουτγάρντι-Ούλμ, ε, για το Παρίσι-Μπρατισλάβα, για αυτή την διαδρομή και στην ε, Στουτγάρδη το 70% ε, των επιβατών μπαίνουν και βγαίνουν και συνεχίζουν όμως μόνο 30%. Αυτή η διαδρομή βέβαια είναι πολύ σημαντική για τις εμπορευματικές μεταφορές. Και από το Παρίσι προς την Πρατισλάβα δεν μπορεί να γίνουν οι εμπορευματικές μεταφορές γιατί η παλιά διαδρομή είναι πάρα πολύ απότομη. Γι' αυτό λοιπόν θα κοστίσουν 3 δις ευρώ, 3 δις μια νέα γραμμή πρόκειται για συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 12 έως 14%. Και ρώτησα, τι γίνεται με αυτή την διαδρομή Εντάξει, ε, είναι ε, κάπως εκεκλημένο έδαφος το, ε, ο σταθμός, αλλά τι θα γίνει με την διαδρομή Και η Κομισιόν μου είπε, αυτή αυτή η διαδρομή με τα 3 δις ευρώ ε, θα είναι ακόμα πιο απότομη. Άρα δηλαδή δεν ταιριάζει για τις εμπορευματικές μεταφορέ. Τι σημαίνουν αυτά εάν οι άνθρωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τόσο χρηματοδότηση και δίνουν 3 δις ε, για αυτή την διαδρομή και για την ε, σύνδεση από τον Περολίνο προς το Ρότσλαφ ή προς άλλες σημαντικές πόλεις δεν υπάρχουν χρήματα αλλά από τη Στουτγάρδη βλέπουμε διάφορες διασυνδέσεις προς την στην ε, Ελβετία πούμε, ή μεταξύ Φράιμπουργκ και Κόλμα και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τα θεωρώ όλα αυτά κοινικά. Το θέμα δεν είναι πόσα χρήματα θα πάρουμε, δεν θα διαγράψουμε τίποτα, γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν θα τελειώσουν ποτέ. Εμεί θα έχουμε πεθάνει και ακόμα αυτοί δεν θα έχουν τελειώσει. Αν μπορείς να απαντήσεις, βεβαίως. <laughs> Θα αφήσω την Επιτροπή να αποφασίσει ποια είναι τα καλά προγράμματα και ποια όχι. Φυσικά αληθεύει ότι όταν ε, βλέπουμε τα κονδύλια από το 2007 ως το 2013 και τα κονδύλια προβλέπονται για το Connecting Europe, συνειδητοποιούμε ότι ε, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, όχι τόσο μεγάλη όπως αυτή που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά ε, είναι μεγάλη αύξηση και υπάρχουν προγράμματα που έχουν περικοπή και αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε αν χρειαζόμαστε όλα τα προγράμματα, ε, γιατί αν είναι όλα εκεί θα έχουν και μικρότερα, μικρότερη χρηματοδότηση. Ε, ή πώς να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα όλα τα χρηματοδοτικά μας μέσα για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εγώ αυτό που φοβόμουν είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ήταν ακόμη πιο αυστηρό για το Connecting Europe. Όμως διατήρησαν αυτή την ε, σημαντική αύξηση. Από την άλλη, όταν εξετάζουμε, όπως είπε και ο κύριος Σερι και άλλους τομείς του προϋπολογισμού, έρευνα παραδείγματο χάρη, άλλο ένα σημαντικό ζήτημα για την Επιτροπή Μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, λέει πώς ε, θα υπάρξει πραγματική ανάπτυξη από το επίπεδο του προϋπολογισμού του 2013. Αν σκάψετε όμως, θα διαπιστώσετε ότι είναι μικρότερη του 5% αυτή η αύξηση. Ε, καταλαβαίνετε ότι δεν, ε, δεν είμαστε και πολύ φιλόδοξοι, ούτε θα χρηματοδοτήσουμε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα με τέτοια αύξηση, με τέτοια αύξηση του 5%. Από το 2007 ως το 2000 13 θα παραμείνουν ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο τα κονδύλια μετά την τελευταία αύξηση. Γι' αυτό είναι αρνητική η έκβαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτό μπορεί να επηρεάσει τους οργανισμούς και άλλες δαπάνες ε, διότι ε, θα κινούμεθα εντός ε, ενός ιδιαίτερα στενού πλαισίου μετά την κατηγορία 1α εάν δεν επιτύχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ή αν δεν τροφοδοτήσουμε την κατηγορία με περισσότερα κονδύλια γιατί ξαναλέω ότι είναι μόνο το 13% του προϋπολογισμού αυτό το τμήμα. Με ρώτησαν πολλοί τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ιζαμπέλ Άιντα. Πολλοί ρωτήσατε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, νέα απάντηση μας δίνει κάθε φορά που θέτουμε το ίδιο ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε την πρότασή της για το πολιτιές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, υπάρχει μια αρχική πρόταση, αλλά έχει ε, τροποποιηθεί σημαντικά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε τις προτεραιότητες και τη διαπραγματευτική εντολή για το Συμβούλιο. Συμφωνία όμως δεν υπάρχει. Είναι ένα εφαλτήριο για τις διαπραγματεύσεις παρόλα αυτά, γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε τέλος. Η γάμα δελτα μπάτς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας είπε ότι κάπου στα μέσα τέλη Μαΐου θα καταθέσουν νέα πρόταση σε αντίθεση με αυτά που μας είχαν υποσχεθεί ότι θα κατέθεταν νέα πρόταση νωρίτερα και ενδεχομένως να, λάβουν, να, λάβει υπόψη η Γενική Διεύθυνση της προτεραιότητας του Συμβουλίου. Ε, θα μπορούσαμε να τους συστήσουμε να εμείνουν στη δική τους την πρόταση και να μην υιοθετήσουν τις γραμμές του Συμβουλίου. Δεν μπορούμε όμως να, να τους το επιβάλλουμε αν δεν το επιθυμούν. Προτείνω λοιπόν, όπως έλεγα, να ε, μείνουμε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα είναι κέριος ο ρόλος Επιτροπής Μεταφορών για τις διαπραγματεύσεις και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του ετησίου προϋπολογισμού, διότι θα ε, συμβάλλει με ιδέες σε σχέση με την προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσουμε για κρίσιμα ζητήματα. Εάν δεν συμφωνήσουμε, αυτό έχει σημασία, αν δεν έχουμε πουδουπού μέχρι το τέλος του 2013 και διατηρήσουμε τα ανώτατα όρια προηγουμένων ετών, τι σημαίνει αυτό, ακόμη λιγότερα κονδύλια για την κατηγορία 1α, για έρευνα δηλαδή, για το συνδέοντα στην Ευρώπη, αλλά όχι, δεν θα μεγάλη μείωση το πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια για τα επόμενα έτη θα δυσκολευτούμε, διότι το ανώτατο όριο το 2013 έχει πολλά κονδύλια για τη γεωργία και ε, αυξημένα κονδύλια για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα έπρεπε όμως να θυμόμαστε εδώ στην Επιτροπή ότι παρά τις περικοπές ε, για το συνδέοντα στην Ευρώπη, αν δεν καταφέρουμε να αυξήσουμε το επίπεδο των κονδυλίων και χρειαστεί να επανέλθουμε, ε, κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε και ο κύριος Κράμερ έχει σχετικές προτάσεις, ε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε να υπάρχει αποδοτικότητα ως προς τη χρήση των κονδυλίων που υπάρχουν. Χαίρομαι που Υπότιτλοι ε, συνεργαστήκαμε αγαστά μέχρι στιγμής και προσβλέπω και στη μελλοντική μας συνεργασία. Ας κάνω και μια τελευταία παρατήρηση. Η Επιτροπή Μεταφορών έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις για να στηρίξει πολιτική μεταφορών και τουρισμού και αυτό φυσικά ε, θα είναι ένα θέμα που θα παρουσιάσει ενδιαφέρον στις διαπραγματεύσεις και όπως σας είπα κάπου το Μάιο, τον Ιούνιο θα χρειαστούμε νέε ιδέε από πλευρά σα. Ευχαριστούμε. Σίμψον. Ευχαριστούμε, Για την παρουσίασή σου και για την απάντηση που έχεις, τις απαντήσεις που έδωσες στα ερωτήματα των μελών. Εγώ συμφωνώ με την Γκεζίνε ότι δεν φαίνεται να είναι η καταλληλότερη στιγμή για να είναι κανείς ε, εισηγητής ή εισηγήτρια του προϋπολογισμού. Είναι όμως σημαντικό να έχουμε συναδέλφους με υψηλή ποιότητα σε αυτό το ρόλο και χαίρομαι που εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών με την κυρία Ντουράν με τους ε, υπόλοιπους σχεδόν εισηγητές μπορούμε να σας δώσουμε πολύ καλή κατεύθυνση για το τι θέλουμε να έχουμε στον τομέα των μεταφορών και ξέρουμε και από την ε, παλαιότερη εμπειρία ότι υπάρχει μία ε, συμπάθεια μεταξύ τη Επιτροπή Μεταφορών και τη Επιτροπή Προπολογισμού. Χαίρομαι για την παρουσία σου και θα τα ξαναπούμε τι επόμενε εβδομάδε. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα τη ημερησία διάταξη που είναι η εξωτερική πολιτική αερομεταφορών τη Ευρωπαϊκή Ένωση έκθεση Μαρινέσκου. Ο κύριος Γκρό θα αντικαταστήσει τον κύριο Μαρινέσκου. Μαθαίε. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ο συνάδελφο κ. σήμερα δεν μπορούσε να έρθει και με παρακάλεσε σύντομα να παρουσιάσω την έκθεσή του. Τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα οι αερομεταφορές ε, να παρουσιάζουν τη θέμενη αξία ύψους περίπου 365 δις. Επίσης ε, θεωρεί ότι στον τομέα των αερομεταφορών απασχολούνται περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη. Ο στόχος μακροπρόθεσμα είναι να βελτιωθούν οι αερομεταφορές ε, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά τώρα τη διεθνή συνεργασία, βεβαίως και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι οι αερομεταφορές, αν δεν λάβει κανείς υπόψη του τη διεθνή διάσταση του θέματος δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν. Ε, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για αερομεταφορές μέσα στην Ευρώπη και σε παρένθεση θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα, το παράδειγμα της ανταλλαγής εκπομπών και κλείνει η παρένθεση. Υπάρχουν λοιπόν οι συμβάσεις που έχουν συναυτεί σε διεθνές επίπεδο, αλλά υπάρχουν και κάποιες συμβάσεις που εκκρεμούν με κάποιες χώρες. Εκεί λοιπόν θα μπορούσαν να συναυτούν επιπρόσθετες συμβάσεις, έτσι ώστε να καλύψουμε αυτή τη διεθνή διάσταση των αερομεταφορών και επίσης ε, μπορούμε να λάβουμε περισσότερο υπόψη μας τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Για μας είναι σημαντικό στον ευρωπαϊκό χώρο να περάσουμε το Single European Sky. Εδώ, κατά την άποψη του συγητή, πρόκειται για δύο σημαντικά θέματα. Πρώτον, η αξιοπιστία της πρωτοβουλίας μας, γιατί εκείνο που επιθυμούμε είναι να επιτύχουμε τη βέλτιστη χρήση αυτού του χώρου. Βέλτιστη χρήση, αυτό σημαίνει και θετικές προεκτάσεις στο περιβάλλον, στην ασφάλεια και γενικότερα στο δυναμικό που έχει η Ευρώπη. Αυτό δηλαδή που έχει και προτείνει η Ευρώπη δυστυχώς πολλές φορές αποτυγχάνει διότι υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη. Και αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό. Ε, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αν η Ευρώπη θέλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Τελευταία παρατήρηση που κάνει ο εισηγητής είναι το εξής. Να υπάρχει στην εργασία και στην ΙΚΑΟ να μην μιλάμε με 27 διαφορετικές αλλά με μία φωνή. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και πέρα από τη θεωρία όλα αυτά να τα μεταφέρουμε και στην πράξη. Κατά τη δική μου λοιπόν την άποψη και αυτό θέλω να το προσθέσω από καθαρά οικονομική σκοπιά οι αερομεταφορές στην Ευρώπη μειώνονται σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Και αυτό φύγει τις αεροπορικές εταιρείες. Άρα δηλαδή πρέπει να τεθεί το ερώτημα σε εμά εδώ πώς ε, αύριο θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα είδη μεταφορών, όπου οι αερομεταφορές είναι και θα παραμείνουν σημαντικές. σημαντικές. Πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη φωνή της Ευρώπης, όχι μόνο από οικονομική σκοπιά, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου ε, Μαρινέσκου και που με παρακάλεσε να σας παρουσιάσω σήμερα σε εσά τους ε, συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε, Ελχαντράου, για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη, διότι δεν μπορεί να έρθει ο ισκιώδης μας. Θα τον... Ε, είναι ο Γιώργο Λάιχτφριντ, θα τον αντικαταστήσω να ευχαριστήσω και εγώ τον ε, κύριο Μαρινέσκου για το σχέδιο έκθεσης. Υπάρχουν ε, διάφορα σημαντικά ζητήματα που ήδη καλύπτονται από την έκθεση. Θα μπορούσε ενδεχομένω να εμβαθύνει σε κάποια άλλα και ως ομάδα θα θέλαμε να προσθέσουμε και εμείς νέα στοιχεία θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην αναθεώρηση των, ε, της οδηγίας για τα δικαιώματα των επιβατών, ε, θεσπίζοντας έτσι το καλύτερο σύστημα παγκοσμίω. Επίσης, να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τις υφιστάμενες και μελλοντικέ οικονομικές προκλήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχυρός ανταγωνισμός, με κάποιες αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής για τις επιδοτήσεις και για τα hubs τους κόμβους. παρακολουθώντας εκ του σε για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στη συνέχεια, ε, η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνισμός για τις τιμές, ντάμπινγκ ε, ε, από ντόπιου αερομεταφορείς, ορισμένες συνθήκες, αθέμητες πρακτικές ως προς τα εργασιακά ζητήματα, επιδοτήσεις για περιφερειακούς αερολιμένες και το καθεξής. Επίσης υπάρχει το θέμα ότι η τωρινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν ήταν και πολύ αποτελεσματική για να καταρτήσει στρατηγικές και να βρει απαντήσεις για διάφορα ζητήματα. Γνωρίζουμε όλο το πακέτο των αερομεταφορών, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνω. Υπάρχει και το στοιχείο ETS, εμπόριο δικαιωμάτων ρήπων, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τομέα των αερομεταφορών τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε βάση σε αυτό το σημείο και έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση, δεν είμαστε σίγουροι, αλλά τουλάχιστον το ελπίζουμε. Στη συνέχεια, ε, τα τέλη για την ασφάλεια στις αερομεταφορές. Ο Γιώργη είναι εισηγητής, όπως γνωρίζετε, και εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία το Μάιο το 2010, με 96% πλειοψηφία και ακόμη παρακολεί τη διαδικασία ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε σχέση τώρα με την ε, κανονιστική σύγκληση. Τι συμβαίνει όταν ανοίγουμε τις αγορές ε, θα πρέπει να ισχύσουν θεμητοί όροι ανταγωνισμού και άρα η ρυθμιστική σύγκληση είναι μία από τις σημαντικότερες πτυχές. Ε, τέλος, μία ενδεχόμενη εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΕΠΑ που επηρεάζει όμως σε μεγάλο βαθμό τον τομέα των αερομεταφορών και ως Επιτροπή Μεταφορών θα έπρεπε να επιληφθούμε και αυτό το σημαντικό ζητήμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίμψον. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ελχαντράουι. Ε, ε, ε, η κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ. Φαίνεται ότι οι συγγητές και οι σκιώδεις απουσιάζουν όλοι, οπότε και εγώ αντικαθιστώ τον σκιώδη μα που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου. που λέει λοιπόν ο σκιώδη μας ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πάρα πολλά σημεία κυρίως ε, το Σίζαρ και τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό ε, και θα ήθελα να προσθέσω ότι το, αν, ε, το ότι δεν προχωρούμε με τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να συμβαίνει αυτό. Ελπίζω να προοδεύσουμε. Τονίζω ο εισηγητή πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ένωση και τι τρίτε χώρε, κυρίω μέσα από διμερεί ε, συμφωνίε και επιθεώρηση των υπηρεσιών των αερομεταφορών. Συμφωνούμε με αυτό, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι οικονομικά επικερδεί αυτέ οι διμερείς συμφωνίε και δεν δημιουργούν πραγματικέ νέε ευκαιρίε για του Ευρωπαίους αερομεταφορεί. Μπορεί να το σχολιάσει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό μα ρωτάει ο κύριος Μπένιεν, για την υποδομή και του κόμβου, ε, τονίζει την ανάγκη τα κράτη-μέλη να είναι ε, πολύ πιο καινοτόμα σε σχέση με τον τρόπο χρήση τη δυναμικότητα των αερολιμένων του. Χρειάζεται ανάπτυξη δευτερογενών των ειδικευμένων κόμβων που εστιάζουν σε, συγκεκριμένους, ε, σε συγκεκριμένες περιφέρειες, ε, τονίζοντας ε, και τη σημασία των περιφερειακών αερολιμένων. Ιδού, λοιπόν, ακούσατε τη φωνή του κύριου Μπένιαν μέσω εμού. Ευχαριστούμε, κυρία Μάισαν, λέει ο κύριο Σίμψον. Η κυρία Μπόστα τώρα. Thank you very, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή κυρία Φώστερ. Ο κύριος Μαρινέσκου έχει δημιουργήσει μια πολύ πλήρη έκθεση. Όπως ε, είπε πολύ σωστά, συζητάμε για αυτά τα θέματα εδώ και πάρα πολύ καιρό και σίγουρα έχουμε πολλές συμφωνίες οι οποίες έχουν συναυτεί σε επίπεδο υπηρεσιών αερομεταφορέων. Είναι καλό το να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιες χώρες όπου πρέπει να πετύχουμε κάποια πρόοδο σε διμερεί γιατί αυτό είναι απαραίτητο για μας. Για την ε, Βραζιλία βέβαια υπάρχουν αυτά τα θέματα για τα οποία συμφωνεί και η Κομισιόν μαζί μου. Για τη γενική του προσέγγιση τώρα. Και πάλι υποστηρίζουμε τη θέση του αυτή για τους ενιαίους ε, εθέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να μιλάμε για τους ενιαίους εθέρες και το σύστημα ΣΕΣΑΡ ως το δυνατόν πιο συχνά υποστηρίζουμε και τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει και αυτά να πιέσουν για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματο και έχει δίκιο η κυρία Μάσνα λέγοντα ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη είναι αποκαρδιωτική και χρειαζόμαστε πιο πολλέ θετικέ ενέργειε για να προχωρήσουμε. Γιατί το σύστημα αυτό δεν περιλαμβάνει την ε, Ιρλανδία και το Ρωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Σκανδιναβία. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τώρα με τη μετάφραση αυτού του εγγράφου στα αγγλικά σε κάποιες παραγράφους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. <clears throat> Απλώς μπορώ να τα επισημάνω αυτά τα σημεία αργότερα. Και άλλα σημεία που έχουν να κάνουν με την αγορά, νομίζω ότι ο κ. Μαρινέσκο έχει μεγάλο δίκιο. Έχει θίξει τα πιο σημαντικά θέματα, το θέμα του ανταγωνισμού με τη Μέση Ανατολή και την Νότια Αμερική και το θέμα του πώς η Νοτιοανατολική Ασία και διάφορα απομακρυσμένα μέρη όπου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τη δημιουργία ικανότητας, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. <clears throat> δεν πρόκειται κανείς να μας αντιμετωπίσει σαν ξεχωριστή οντότητα την Ευρώπη, γιατί έτσι δουλεύει ο κόσμος. Θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε, να κατανοήσουμε ότι ο κόσμος προχωράει. Σε κάποια μέρη του κόσμου οι αερομεταφορείς ενισχύονται, και εμείς θα πρέπει να έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση ώστε οι δικές μας εταιρείες να εξασφαλίσουν θεμητό ανταγωνισμό μαζί τους και να έχουν μια διεθνή παρουσία στο βαθμό του δυνατού. Και τέλος, οι προτάσεις του κ. Μαρινέσκο για τις μελλοντικές δράσεις θίγουν σημαντικά σημεία, ιδίως το θέμα για τις αθέμητες τιμολογικέ πρακτικές και το γεγονός ότι υπάρχουν αερομεταφορείς τρίτων χωρών που υποστηρίζονται από τι κυβερνήσει του. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η δική μα πολιτική όμω είναι σαφής ότι θα υπάρχει επιχορήγηση προ του ε, αερομεταφορεί. και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε καλή κατάσταση ανταγωνισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Χωρί φυσικά να μπορούμε να επηρεάσουμε τι κάνουν οι άλλε τρίτε χώρε. Ο Σάιντ μίλησε για το σύστημα ITS για την εμπορία εκπομπών. Στην παράγραφο 32 όμως, ίσως πρέπει να τα πούμε αυτά πιο σαφώς, αλλά αναφέρθηκε και ο ρόλος της ΙΚΑΟ και τα μέτρα που βασίζονται στην αγορά και ίσως εκεί μπορούμε να έχουμε μια λύση για τα θέματα του ETS, αν και αμφιβάλλω. Αν θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, θα γίνει κάτι τέτοιο. Εξ ονόματος του συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ευχαριστούμε τον κύριο Μαρινέσκο και θα έχει την υποστήριξή μας στη συνέχεια της επεξεργασίας της έκθεσης αυτής. Λάχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ για την ε, έκθεση. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα ε, που θα ήθελα είτε να τα ενισχύσω είτε να προσθέσω ε, κάποια σημεία. Βεβαίως, ε, λόγω της ε, κατάστασης ε, που συζητήσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εμπορία εκπομπών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα σε αυτή την έκθεση και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την εμπορία των εκπομπών. Να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις τους σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι πέρα από την εμπορία εκπομπών πρέπει να θίξουμε και το θέμα του θορύβου. Ε, και στα αεροσκάφη υπάρχει διαφορετική ποιότητα θορύβου και όταν όλα αυτά τα αεροσκάφη έρχονται στην Ευρώπη πρέπει να σας πω ότι δημιουργούν πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι εντωμεταξύ υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με το διοξίδιο του άνθρακα αλλά και με το οξύδιο του αζότου. Και υπάρχουν υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται όλο και πιο ουσιαστική σχετικά με τις ε, εκπομπές ε, στην ε, υψηλή σφαίρα, σε υψηλά επίπεδα της στρατόσφαιρας, που νομίζω ότι ε, λόγω της αυξανόμενης ε, ποσότητά τους ε, αυτά δεν πρέπει να τα αγνοούμε. Και αυτό πρέπει να το θίξουμε σε διεθνές επίπεδο, γιατί αυτό δεν σημαίνει μόνο σε εμά, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Συμφωνώ λοιπόν με τον συνάδελφό μου από τους σοσιαλδημοκράτες, ότι και το θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών και αυτό πρέπει να το προβάλλουμε περισσότερο. Διότι θεωρώ ότι στο θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών θα πρέπει να υιοθετηθεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα δηλαδή εμείς να μην αποδυναμώσουμε τα δικαιώματα αυτά γιατί μπορεί να συμβεί το εξή. Ναι, μεν θεωρητικά να μην μειωθούν τα δικαιώματα, αλλά να έρονται επί της ουσίας όταν προκύπτει μια μεγάλη καταστροφή. Δεν πρέπει να συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Και κατά την άποψή μου πρέπει να αμφισβητήσουμε λιγάκι ε, τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφεί για αυτό το θέμα. Όσον αφορά το Single Sky, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα αξιοπιστίας αν έχουμε μόνο κάποια τμήματα του ε, εναέρου χώρου όπου λειτουργούν τα πράγματα και ρυθμίζονται κανονικά. Και κατά τα άλλα υπάρχουν ε, μόνο δηλώσεις προθέσεων. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι στην Κομισιόν να μην μιλάει για τμήματα συγκεκριμένα του εναέρου χώρου, να μιλάει ότι εδώ πρόκειται για κάποιο πρώτο βήμα ε, και με το γεγονός ότι θα υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία, κατ' ουσίαν δεν θα αλλάξει τίποτα. Όσον αφορά τώρα τις ε, κρατικές επιχορηγήσεις, νομίζω ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην Ευρώπη τρέχουν αρκετές ε, διαδικασίες επί παραβάση, ε, επιχορηγήθηκαν παράτυπα πολλά αεροδρόμια από διάφορα κράτη-μέλη και γι' αυτό λοιπόν πρέπει, εφόσον επιθυμούμε να λειτουργούν σωστά τα αεροδρόμια, ε, να διοργανωθούμε κατά πόσο συμβαίνει σε αυτή πρόκειται για συγκαλυμμένες επιδοτήσεις. Κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα σας πω ένα νεκροτάκι τώρα, μία μικρή ιστοριούλα. Έχουμε τρία άτομα τρία μικρά γουρουνάκια συγκεκριμένα. Ένα έχει ένα αχυρένιο σπίτι, το άλλο ξύλινο σπίτι, το άλλο τούβλινο σπίτι. Το πρώτο μικρό γουρουνάκι λοιπόν είναι η βιομηχανία. Η αεροναυπηγική βιομηχανία της Ευρώπης που έχει ενωθεί για να φτιάξει ένα ενιαίο φορέα και φυσικά υπάρχει μεγάλη επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πουλήθηκαν 200 αεροπλάνα το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το γουρουνάκι που έχει το ισχυρό το τούβλινο σπίτι. Το δεύτερο είναι οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, ενώνονται, συγχωνεύονται, εξαφανίζονται, έχουν λύματα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως τα καταφέρουν και μαζί τους τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν και αυτά πολλές δυσκολίες και επαναδιοργανώσεις. Αυτό είναι το γουρουνάκι που έχει το ξύλινο σπίτι και μετά έρχεται η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση η οποία δεν μπορεί να έχει κάτι καλύτερο από ένα χειρένιο σπίτι. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε, να διορθώσουμε σωστά τον εναέριο χώρο της Ευρώπης. Η, ενα, η ενιαία είναι σε κατάσταση ικτρή, το ΣΕΖΑΝ σε κατάσταση ικτρό ικτρή, η διαλειτουργικότητα επίσης και μια δεύτερη τώρα πτυχή που πρέπει να θίξω είναι το θέμα των, του ρυθμιστικού πλαισίου μέσα στην, ε, στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο καθορίζουμε ορισμένα θέματα που είναι το πλαίσιο, το περιβαλλοντικό, το κοινωνικό, δικαιώματα των επιβατών, τα θέματα ασφαλείας κτλ. Εκεί προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο. Να έχουμε το πιο απαιτητικό πλαίσιο, το οποίο θα εξασφαλίσει και στον επιβάτη και στον εργαζόμενο την ασφάλειά του, την ποιότητα κτλ. Και θα βοηθήσει όλη την οικονομία της Ευρώπης. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι <clears throat> το σύστημα αυτό έχει ένα διεθνή χαρακτήρα. Η όλη αεροπορική βιομηχανία και όταν θέλουμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό έρχεται ο Λύκος και λέει στα γουρουνάκια έλα εδώ, έλα εδώ. Και εκεί αντιμετωπίζουμε λοιπόν τα προβλήματα του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των επιβατών, την ε, ηχορύπανση, τα θέματα ασφαλείας, όλα αυτά λοιπόν τα ρυθμίσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μετά πρέπει να κάνουμε και κάποιε συμφωνίε με του διεθνεί εταίρου μα για τα θέματα αυτά και δεν έχουμε καμιά δυνατότητα να προστατευτούμε από τον λύκον. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν έχουν διεθνή χαρακτήρα. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω τα κράτη-μέλη να μπορούν να πάνε να κρυφτούν στο σπίτι από τούβλα που έχει φτιάξει η αεροπορική βιομηχανία αλλά στα άλλα σπίτια δεν έχει πραγματική προστασία. Έχουμε όλους τους εργαζόμενους που έχουν να αντιμετωπίσουν συνεχείς αναδιαθρώσεις που οδηγούν πολλές φορές σε απόλυση. Έχουμε τα προβλήματα του περιβάντος που έχουμε όλο και μεγαλύτερη δυσκολία για το σύστημα παραγωγής χάρη εμπορίας εκπομπών και επομένως η διάκριση μεταξύ ενός ιδεατού πλαισίου ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αερομεταφορές και της ανάγκης να λειτουργήσει σε διεθνές πλαίσιο όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σχιζοφρενικό. Αυτό ήθελα να σας πω. Thank you very much, Σα Σας ευχαριστώ. Αν ποτέ αποσυρθείτε από τον πολιτικό βίο, θα κάνετε πολύ καλή καριέρα ως ε, συγγραφέας ε, ή μάλλον ε, παρουσιαστής παιδικών εκπομπών στη γαλλική τηλεόραση. Ο Λύκος είναι το συμβούλιο μας, είπατε, προσπαθεί φυσώντας να καταστρέψει τα χειρένια σπιτάκια. Πολύ μ' άρεσε αυτό. Κύριος Μπάχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα το να το παρουσιάσει κανείς ε, τόσο ε, γλαφυρά και με τέτοιο χιούμορ όπως το έκανε ο συνάδελφός μου, εγώ σίγουρα δεν θα τα καταφέρω. Και θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Μαρινέσκου γιατί παρουσίασε μια πολύ καλή έκθεση και τα σημαντικότερα θέματα όχι μόνο τα έθιξε, αλλά κατέθεσε και σχετικές προτάσεις. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι στόχοι, παρότι επιτεύχθηκε πρόοδος, τελικά δεν έχουν επιτευχθεί. Και υπάρχει ένα θέμα το οποίο θέλω να αναφέρω. Το περισσότερη Ευρώπη. Ε, Παρότι, παρότι λοιπόν ε, στο προηγούμενο θέμα ε, της ε, επίγειας εξυπηρέτησης τάσσομαι υπέρ της επικουρικότητας, Όσον αφορά όμως στις αεροπορικές μεταφορές, εκεί πρέπει να έχουμε περισσότερο ενιαίες, μια ενιαία πολιτική, να έχουμε θεμητό και δίκαιο ανταγωνισμό, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην έχουν αντιμετωπίσει να θέμει τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Να είναι σαφείς οι προδιαγραφές ε, ε, οι προδιαγραφές για το περιβάλλον, τα δικαιώματα των επιβατών. Υπάρχουν ευρωπαϊκές ε, ε, προδιαγραφές που επιτρέπουν τον θεμητό ανταγωνισμό. Ως εισηγητής στην Επιτροπή Απασχόλησης προφανώς και θα δώσω μεγαλύτερη σημασία στις προϋποθέσεις απασχόλησης και ελπίζω να με στηρίξει η Επιτροπή Μεταφορών. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπάλντον, πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς ποιο, σπιτάκι θα φυσήξετε για να <laughs> πέσει. Ε, πρόεδρε, δεν είμαι σίγουρο και πρέπει να βρω και εγώ μια παιδική ιστορία για να απαντήσω. Λοιπόν, δυστυχώ δεν μπορώ να συμβάλλω και τόσο πολλά σε αυτή την τόσο χρήσιμη συζήτηση. Ευχαριστούμε για τον εισηγητή, για το σχέδιο έκθεση. Ε, καλύπτει ικανοποιητικά το ζήτημα πιστεύουμε και μα ικανοποιεί διότι ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση με τη δική μα ε, ανακοίνωση και τα συμπεράσματα του Σύμβουλου. Υπάρχει δηλαδή ομοψυχία σχετικά με το τι πρέπει να γίνει. Ε, θα μπορούσα να σχολιάσω πολλά επιμέρου σημεία, αλλά δεν είναι η δική μου δουλειά. Θα σα πω ότι για τον ενίο Ευρωπαϊκό Ουρανό συμφωνούμε. Συμφωνούμε με τα σχόλια για τη Βραζιλία, για τον κόλπο και τα κράτη του. Και φυσικά το ζήτημα τη εμπορία εκπομπών πρέπει να μα απασχολήσει στο μέλλον. Υπάρχουν δύο ουσιαστικά ζητήματα που θα ήθελα να σχολιάσω περισσότερο. Ο κύριο Ελχαντράβη μα μίλησε για την εμπορική συμφωνία ΕΕ και την προσθέμενη αξία που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αν συμβάλλουμε ικανοποιητικά. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι εξελίξει. Πρώτη φορά θα συζητηθεί το θέμα ελευθέρων εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στην Ένωση και τη ΙΠΑΕ και θα έπρεπε η αεροπλοεία να έχει ένα σημαντικό ρόλο ε, στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων. Δεν θα πρέπει να επιμείνουμε για τα ζητήματα ιδιοκτησία και άλλα που είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα, αλλά μπορούμε να έχουμε μια θετική συμβολή και ξαναλέω να φέρουμε προσθέμενη αξία όσο προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Δεύτερο σημείο ίσω να είναι και ζήτημα μετάφρασης. Ε, μας είπε η, Foster, η κυρία Φώστερ ότι υπάρχει το σημείο 30, λέει η έκθεση, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνάψει μια δίκαιη συμφωνία με τη Ρουσική Ομοσπονδία για τις ε, ε, υπερσιβηρικές οδούς και την υφιστάμενη συμφωνία. ακόμη και, δηλαδή, ο Χάλς Κρίστιαν δεν θα μπορούσε καν να σκεφτεί να παραμύθι για αυτό το ζήτημα ακόμη και αν έγραφε χρόνια. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις υπερπτήσεις πάνω από τη Σιβηρία ε, ε, δεν ήταν, ε, ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Μήπως θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε να, υπάρχει, να υπάρχουν αμοιβαίως παραχωρήσεις για το θέμα των των υπερπτήσεων πάνω από την ε, Σιβηρία. Θα ήταν πιο ήπια η διατύπωση. Ε, ο κύριος Σίμψον, σας ευχαριστούμε κύριε Μπάλτουεν. Ε, κύριε Γκαρσία, έχετε κάτι να προσθέσετε σε σχέση με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Όχι, απλώς μπορώ να προτείνω στον Ντόμινικ να γράψει ένα βιβλίο «Η Ευρώπη όπω τη διηγούμε στα μικρά, στα μικρά παιδιά». Θα ήταν πολύ θετικό και φυσικά θα αναφέρω στον κύριο Μαϊνέσκου τη δασκόλη του κύριου Χέντεχ. Και επίσης για την, ε, τις, τις, ε, τα σχόλια που έγιναν για τη διατύπωση και <clears throat> θεωρώ μετά από αυτά που άκουσα ότι είναι μια καλή έκθεση και αποκομίζει τη γενική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι προθεσμία για τις τροπολογίες 27 Μαρτίου το μεσημέρι 22-23 Απριλίου θα εξετάσουμε αυτές τις ε, τροπολογίες και θα ψηφίσουμε σε 7 Μαΐου στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, 27 Μαρτίου, καταληκτική προθεσμία. Έχουμε εξαντλήσει την ημερησία διάταξη για σέμα. Ξεκινάμε τώρα τη συνάντηση των συντονιστών. Αν θέλετε να φύγετε λοιπόν, μπορείτε να φύγετε. μας διώξουν. Five minutes, coordinators. Σε πέντε λεπτά συνεδριάζουν οι συντονιστές.